Συνεχίζει τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης με τα έγγραφα που έχουν εγκριθεί είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Εγκρίνονται.